δική μου γλώσσα. ξεκινήσω λοιπόν. Αξιότιμα. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι συμμετέχοντες, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ σήμερα στην Διεθνή Μέρα της γυναίκας. Εκπροσώπους 15 κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και, ιδιαίτερως θέλω να καλωσορίσω, ε, τους και τις εκπροσώπους από χώρες υποψήφιες. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε με χαρά να χαιρετήσουμε την παρουσία και εκπροσώπων κοινοβουλίων των χωρών της γειτονίας, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Τινησία και Μαρόκο. Χαίρομαι λοιπόν είστε εδώ σήμερα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε πριν μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, παρεμβάσεις και τη συμβολή στη συζήτηση. Το θέμα μας λοιπόν είναι η οικονομική χειραφέτηση της γυναίκας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε τη διερμηνία σε όλες σχεδόν τις, Ευρωπαϊ... Ε, τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Μαλτεζικής, Λετωνικής και Εσθονική. Επιπλέον δε αυτών έχουμε πέντε γλώσσες που δεν ανήκουν σε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλβανική, αραβική, μακεδονίτικη, τουρκική, ρωσική και παθητικά έχουμε σερβικά, βοσνιακά και μαυροβουνιακά. Υπενθυμίζω ότι η σημερινή μας συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένων και των workshop μεταδίδεται ολόκληρη μέσω του διαδικτύου, ζωντανή. Ε, κατά τη διάρκεια αυτής της εναρκτήριας εκδήλωσης δεν θα μπορέσουν όλοι να μιλήσουν βέβαια, αλλά θα έχετε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των workshop. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Αντώνιο Ταγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, χωρίς παρατέρα καθυστέρηση σας δίνω τον λόγο. Euh, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Γυναικών, κυρία Επίτροπε Γιούροβα, αγαπητοί εκπρόσωποι ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα των γυναικών, αγαπητοί Γενική Γραμματεύ της Οργάνωσης της Γαλλοφωνίας, κυρία Ζαν, και δόκτωρ Σίβα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να κηρύξω την έναρξη της έκτακτης αυτής της συνεδρίασης της Επιτροπής Γυναικών. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη προσέλευση με την ευκαιρία της επαιτίου της Παγκόσμιας Μέρας των γυναικών. Προφανώς είναι μια εκδήλωση εορτασμού. Αλλά δεν πρέπει να έχει μονάχα ρητορικό χαρακτήρα αυτή η εκδήλωση. Γιατί όσο οι γυναίκες είναι θύματα βίας, διακρίσεων, ακροτηριασμών, υποχρεωτικών γάμων. Όσο αποκλείονται από την παιδεία, από τον κόσμο της εργασίας, από την οικονομία, από την πολιτική, από θέσεις ευθύνε. Εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε 365 μέρες το χρόνο για να μπορέσουμε να τονίσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού τον, την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Την τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, τους πολέμους, την ένδια, την ανεργία χωρίς να υπάρξει μια πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών. Μόνο αν δώσουμε πραγματικά στις γυναίκες τη δυνατότητα να εκφραστούν πλήρως σε όλους τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας που θα έχουμε ένα κόσμο πιο ασφαλή, πιο δίκαιο και πιο ευμαρή. Το θέμα της, ε, το, αυτού του χρόνου είναι το οποίο θα μας απασχολήσει είναι οι δυνατότητες της γυναίκας στον οικονομικό στίβο. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία της Μισελ Ζάνι, η οποία είναι Γενικός Γραμματέας της, οργάνωσης για, της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Γαλλοφωνία, με την οποία <clears throat> θα έχω την δυνατότητα να έχω επαφή αργότερα, για το σημαντικό ρόλο που παίζει η Γαλλοφωνία για το θέμα αυτό. Και επίσης για την ιδίω για την προώθηση του επιχειρήματος μεταξύ των γυναικών στην υποσαχάρια γαλλόφωνη Αφρική. <clears throat> Όπως ξέρετε υπήρξε Ευρωπαίος Επίτροπο για τα θέματα βιομηχανίας και του επιχειρήν και αυτό ήταν και μία από, τις, από τους πυλώνες κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Συνεχίζω στα Ιταλικά. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απονείμει το πιο το βραβείο με το μεγαλύτερο κύρος που απονέμει, το βραβείο Ζαχάροφ, σε γυναίκες θαραλέες που ενσωματώνουν ε, αγώνες για τα δικαιώματά τους. Η παραδείγμα στη 16χρονη Πακιστανή Μαλάλα Γιουφσαφσάη η οποία κατέστη σύμβολο του αγώνα κατά της, ε, της, ε, των θρησκευτικών εξτρεμισμών όταν ε, υπέστη επίθεση από τα Λιμπάν βγαίνοντας από το σχολείο της στην Άντια Μουράν και τη Μάχα Μαχαζιμπασάρ από την Εθνικό Θρησκευτική Μειονότητα των Γεζιντή τουρκόφωνες, ε, κουρδόφωνες, συγγνώμη, την οι οποίες έπεσαν θύματα διωγμών από το ΙΣΙΣ. Επίσης ε, συνάντησα πρόσφατα και τη Λαϊμα Μπασάρ και την ε, Νιγηριανή δικηγόρο των δικαιωμάτων και εκείνη έχει θυμηθεί με το βραβείο Ζαχάβροφ, τη Χάουβα Ιμπραήμ. Και οι δύο είναι εδώ παρούσες στην ημέρα της γυναίκας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ το θάρρος τους. Θέλω επίσης όμως να υπενθυμίσω την Ναμίγα Ζιατέν, μητέρα του Γάλλου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του πέρσι στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας μιλήσει για το ρόλο των γυναικών μουσουλμανίδων κατά της ε, θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης. Μητέρα, μουσουλμάνα, μουσουλμάνου στρατιώτου που οι οι τάχα αγωνιζόμενοι στο όνομα του Ισλάμ φώνευσαν. Πώς μπορεί μια γυναίκα λοιπόν να είναι το υπόδειγμα και να ε, μεγαλώσει τα παιδιά της με το πνεύμα του ανοίγματο και της διακλακτικότητας όταν η ίδια είναι στο περιθώριο, όταν αποκλείεται από την παιδεία, από την εκπαίδευση, ε, από την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Είναι πολλές οι συγκρούσεις, οι καταχρήσεις, οι ακρότητες που μπορεί να ξεκινούν από τον φόβο των ανδρών για το δυναμικό των γυναικών. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να μιλούμε μόνο για τη βία, γιατί αυτή η βία ε, σημαίνει και κακομεταχείριση, ταπείνωση μέσα και στην οικογένεια ακόμη του ρόλου της γυναίκας. Και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το παράδειγμα. Γι' αυτό ζητούμε μια κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και των θεσμικών οργανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κύρωση της Σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών και της συνδοοικογενειακής βίας. Είμαι υπερήφανος που είμαι πρόεδρος ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός θεσμικού οργάνου που κάθε μέρα ύψουν τη φωνή του ξεκάθαρα για τα δικαιώματα των γυναικών. Το Κοινοβούλιο προάγει τα δικαιώματα αυτά σε κάθε σχετική απόφαση. Υπάρχει Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διαρκώς εργάζεται για την ισότητα μεταχείριση των φύλων και για τα άλλα δικαιώματα των γυναικών. Αλλά για να περάσω τώρα στο θέμα του ρόλου των γυναικών στην οικονομία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όλοι οι δείκτε δείχνουν πω όσο πιο μεγάλο είναι ο ρόλο αυτό των γυναικών, τόσο μεγαλύτερη και η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση. Οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες μάνατσερ κερδίζουν και σε αποτελεσματικότητα και σε αποδοτικότητα. Ε, το να μπαίνουν στο περιθώριο λοιπόν της οικονομίας οι γυναίκες έχει τεράστιο κόστος, 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, λιγότερη ανάπτυξη μέχρι το 2025 που σημαίνει ΑΕΠ της Ιαπωνίας, Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί. Για σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Πολλά ακόμα έχουμε να κάνουμε. Μόνο το 24% των στελεχών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γυναίκες και μόλις το 4,6% έχουν ρόλους διευθυντικών στελεχών. 655 εκατομμύρια γυναίκες εργάζονται λιγότερες δηλαδή, 655 εκατομμύρια γυναίκες, λιγότερες εργαζόμενες από ό,τι αντίστοιχα οι άντρες. Ο 88% των γυναικών σε ηλικία μεταξύ 30 και 39 ετών διαπιστώνουν ότι με, την, ε, με το να δώσουν ζωή στα παιδιά τους χάνουν και εισόδημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι στην πρώτη γραμμή στο μέτωπο αυτό. Η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια στις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ε, ενταγμένες στα χρηματιστήρια ε, διαρκώς αυξάνεται, διπλασιάζεται από το 11,9 το 2010 έχει περάσει το 22,7 το 2015 αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει αρκετά. Δεν υπάρχει επαρκής ε, εκπροσώπηση και βεβαίως υπάρχει μεγάλη διαφορά και στους μισθούς που φτάνει και στο 16% ακόμη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει στην πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των κοινωνικών στα συμβούλια, διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Ζητούμε επίσης ευρωπαϊκή νομοθεσία σύγχρονη με μεταρρύθμιση της άδειας μητρότητας πέραν των παραδοσιακών ρόλων και τη άδικη κατανομή των καθηκόντων. Εργαζόμαστε για να προαγάγουμε την ε, απελευθέρωση, την οικονομική, τη χειραφέτηση τη γυναίκα και να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές και στους, ε, στα επίπεδα των συντάξεων και των συντάξεων που χορηγούνται ανάλογα του γένους, του φύλου. Θέλουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν προέδρους επιτροπών με ισότιμη εκπροσώπηση, 12 άνδρες, 12 γυναίκες και στο δικό μου βεβαίω το επιταλείο έχουμε ρημνήσει για την ίδια ισορροπία. Και όμως δυστυχώς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικές ημέρες είδαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο να εκτελήσεται. Ένας βουλευτής προσέβαλε κατά τρόπο απαράδεκτο την ισότητα των φύλων απεύθυνε ε, προσβολές προς όλες τις γυναίκες, παραβιάζοντας θεμελιώδες μας αξίες. Δεν σκοπεύω να ανεχθώ τέτοια συμπεριφορά. Ακόμη δε πιο σοβαρή, καθώς εκφράστηκε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, εκεί που θα έπρεπε με αξιοπρέπεια να εκπροσωπούνται όλοι οι ευρωπαϊκοί ε, λαοί. Και έχω αμέσως ζητήσει την ε, κίνηση μιας έρευνας στην οποία σκοπεύω να δώσω άμεσα, το δυνατόν πιο γρήγορα δηλαδή, τις ε, σχετικές κυρώσεις, ανάλογα με, ανάλογες με τη σοβαρότητα αυτών των δηλώσεων. Στα αγγλικά. Κυρίες και κύριοι, κάποια από τα κράτη-μέλη έχουν καλή εμπειρία ως προς την ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Άλλες χώρες έχουν καλά καθεστώτα για την προστασία της μητρότητας ή μπορούν να προσελκύσουν περισσότερες γυναίκες στον χώρο της επιστήμης. Πρέπει να χαιρετήσουμε σήμερα τη συμβολή των γυναικών στις οικονομίες μας και επίσης να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κερδίσουμε σε πρόοδο διδασκόμενοι ο ένας από τον άλλον. Πρέπει να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να προχωρήσουμε μαζί στη χειραφέτηση των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης καθοδηγείται από την προσήλωσή της στις αρχές της ισότητας και στις εξωτερικές της δράσεις. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει αντιπροσωπεία στην ετήσια Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών και τη Επιτροπή για το Καθεστώ των Γυναικών για να συναντηθούν με αντιπροσωπείς από όλο τον κόσμο. Φέτος λοιπόν το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη ήταν η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών σε έναν ε, μεταλλασσόμενο κόσμο εργασία. Το Κοινοβούλιο ιδιαίτερη σημασία μάλιστα αποδίδει στη συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα στι χώρε υποψήφιε, στι χώρε προσχώρηση και στην ευρωπαϊκή γειτονία. Καλωσορίζουμε λοιπόν του εκπροσώπου των κρατών αυτών εδώ και ελπίζουμε ότι η συμμετοχή του στη συζήτηση θα εντείνει και τη συνεργασία μα στον τομέα αυτό. Επίσης θα θέλαμε ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε τη σημαντική έκθεση της Ένωσης ε, των Διεθνών Μουσείων Γυναικών και την ε, παρουσία του Επιτρόπου Κάρλος Μοέδας ε, με την και των γυναικών προσκεκλημένων στην εκδήλωση αυτή σήμερα το βράδυ. Ωστόσο και μετά όλες όλους τους αγώνες για την ισότητα έχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Και έτσι σταματώ για να περάσω στα ισπανικά, είναι απαραίτητο να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα εγχείρημα που εμπλέκει όλους τους βουλευτές και όλες τις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για αυτό το λόγο, για μας, η Ευρώπη δεν είναι μονάχα το ευρώ, <clears throat> δεν είναι μονάχα η κεντρική τράπεζα. Είναι και οι αξίες που συμμεριζόμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο <clears throat> να υπερασπιστούμε όλες τις αξίες και τις αρχές μας και αυτό περιλαμβάνει την αξιοπρέπεια και την ισότητα των γυναικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θερμά για την ομιλία σας για το γεγονό ότι επαναλάβεται ότι μεταξύ των αξιών και των προτεραιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου είναι η ισότητα των φίλων. Στου κόλπου του Κοινοβουλίου ουδέποτε μπορούμε να ανεχτούμε να ταπεινώνονται οι γυναίκε, να υποβαθμίζονται και δεν μπορούμε να το δεχτούμε από την πλευρά οποιοδήποτε μέλο του Κοινοβουλίου, όπω την περασμένη εβδομάδα με το παράδεκτο συμβάν. Να προχωρήσουμε. και είναι μεγάλη μου χαρά να καλωσορίζω την Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα, που είναι υπεύθυνη για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή μας, η Επιτροπή των Γυναικών, έχει πολύ στενή συνεργασία μαζί της. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Ζαν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες ε, και όλους εσάς που ήρθατε από όλη την Ευρώπη σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Είναι μια σημαντική μέρα για μένα, για τις γυναίκες, αλλά ε, υποθέτω και ελπίζω και για τους άντρες. Είναι ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μας, αλλά να κάνουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Να σταθμίσουμε και να αξιολογήσουμε το που έχουμε φτάσει στην Ευρώπη, τι έχουμε πετύχει και τι απομένει να γίνει ακόμη. Σήμερα δημοσιεύσαμε αυτή τη νέα προσθήκη, θα έλεγα, στην ετήσια έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εδώ βλέπουμε ότι πρόοδος έχει επιτευχθεί κυρίως στην αγορά εργασίας, στην απασχόληση των γυναικών, που φτάνει σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, 65, σε ένα ρεκόρ μάλλον του 65,5% και βάσει των στοιχείων της, του Eurostat το μισθολογικό χάσμα ε, έχει φτάσει 16,3% το 2016 από 16,7% τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο μας επίτευγμα. Ε, πρέπει να πετύχουμε περισσότερη πρόοδο και περισσότερο βάσιμη και πιστική. Προλίγου σήμερα είχα μία ακόμη θετική εμπειρία. Βρέθηκα σε μια συνέντευξη τύπου στους χώρους της Επιτροπής με καταπληκτικές κυρίες να συμμετέχουν. Κυρίες που χάρη στα πολύ ισχυρά κίνητρά του, ε, μία από το χώρο των επιχειρήσεων, μια άλλη από ένα think tank και μια ε, αγωνίστρια κατά του ακροτεριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων, ε, όλες μαζί συμφωνήσαμε ότι εμείς που πετύχαμε, είμαστε πετυχημένες πιστεύω γυναίκες, όλες εδώ σήμερα, ε, συμφωνήσαμε ότι είναι καθήκον μας να κάνουμε πολύ περισσότερα για όσες και όσους χρειάζονται βοήθεια. Και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες που είναι δυνατές, είναι ισχυρές, να δυναμώσουν κι άλλο είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, αλλά και εκείνων που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Να αναφέρω μόνο τρεις ομάδες γυναικών. Θύματα βίας, είναι πολύ υψηλή η αριθμή εδώ. Είναι πολλές οι γυναίκες που υποφέρουν και ελπίζουν ότι θα τους στείλουμε χείρα βοηθείας. Να αναφέρω τις γυναίκες της που είναι μόνες και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά ε, για να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες στην Ευρώπη. Θα γνωρίζετε ότι το κλίμα στις κοινωνίες μας υποβαθμίζεται, επιδεινώνεται. Οι επιθέσεις κατά των γυναικών ε, πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη. Βλέπουμε να υπάρχει έλλειψη ανεκτικότητας εις βάρος των γυναικών και ακούμε απίστευτες δηλώσεις Είμαι πραγματικά ευγνώμων, κύριε Πρόεδρε, και σε εσά και στο Ευρωκοινοβούλιο για την πολύ άμεση και σταθερή δράση που αναλάβατε κατά του μέλους του Κοινοβουλίου και του απίστευτου συμβάντος που προκάλεσε στην Ολομέλεια την περσμένη εβδομάδα. Βλέπουμε ότι οι προκαταλήψεις κατά των γυναικών εμένουν Πρέπει να δράσουμε λοιπόν. Βάσει του Ευρωβαρόμετρου για την βία κατά των γυναικών, 70% των γυναικών στην Ευρώπη ε, αναφέρουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι το σύνηθε στις χώρες τους. Η βία λοιπόν εις βάρος των γυναικών και η εκστρατεία που οργανώνουμε φέτος με πολύ καλή χρηματοδότηση είναι μια εκστρατεία στην οποία θα ευχαριστούμε τη βοήθειά σας. Θέλουμε τη συμμετοχή σας για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Εμένουν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω χάρη ε, ότι η ενδοκοκενειακή βία είναι κάτι το κανονικό, το ομαλό. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Η βία κατά των γυναικών υπονοεί ότι, πρέπει, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ένοχη συμπεριφορά και από την πλευρά του θύματο. Αυτό πρέπει να ανατραπεί στην Ευρώπη. Για το μισθολογικό χάσμα, αναφέρατε και εσεί του αριθμού, ε, Πρόεδρε. 16,3% το 2016 και για τις συντάξεις μιλάμε για 38%. Για μένα αυτό είναι πραγματικά ένα στοιχείο που θα έπρεπε να μας ε, προκαλεί ενοχές. Δεν κάνουμε αρκετά για μένα το να έχουν τόσο, χαμηλές, τόσο χαμηλές οδήματα οι ηλικιωμένες γυναίκες είναι ντροπή. Ντροπή για την κοινωνία μας. Είναι ντροπή για γυναίκες που δούλεψαν όλη τους τη ζωή και μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Επίσης η περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Μία στις 20 διευθύντρες εταιριών είναι γυναίκες ε, στην Ευρώπη. αλλά αν 60% ε, των πτυχιούχων ε, των ε, πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων είναι γυναίκες, πού εξαφανίζονται στην πορεία. Πώς δεν γίνονται διευθύντριες. Πρέπει κάτι να κάνουμε και γι' αυτό. Ε, Μιλώντα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πω ότι συνεχίζουμε να πιέζουμε για βελτιώσει, χρησιμοποιώντα όλα τα απαραίτητα μέτρα, είτε είναι νομοθετικά αυτά, είτε μη νομοθετικά και σχετικέ δράσει μη νομοθετικέ. Συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράση και εντό Ευρώπη και εκτό, και θέλω να αναφέρω κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, αφιέρωσε το 2017 στην εκρίζωση κάθε μορφή βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Να θυμίσω εδώ, Πρόεδρε, την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Θα πρέπει να πιέσουμε τα κάτι μελη που δεν έχουν κυρώσει αυτή την ε, σύμβαση να το κάνουν άμεσα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα ώστε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Θα πρέπει να γίνει αυτό αμέσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο θα υποβάλει μια πρωτοβουλία για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου για του γονεί και του φροντιστέ στι 26 Απριλίου κανονικά φέτο ε, και υπολογίζω στη στήριξή σα, τι αντιδράσει και τα σχόλιά σα μετά από ευρύτατε διαβουλεύσει που έχουμε διοργανώσει και νομίζω ότι θα πετύχουμε να, πε... να συνθέσουμε ένα, μια δέσμη μέτρων νομοθετικών και μη νομοθετικών που πολύ σύντομα θα μας φέρουν θετικά αποτελέσματα. Επίσης, προτείναμε αλλαγές στη μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου για να προστατεύονται καλύτερα οι γυναίκες μετανάστευες που φτάνουν στην Ευρώπη. Επίση, υποστηρίζουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και τον οικογενειακό σχεδιασμό με τις σχετικέ υπηρεσίες. Στα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν και τις όλες συζητήσει. Α ε, ενσκύψουμε σε αυτά τα τόσο ε, συναρπαστικά ζητήματα, να μάθουμε ημένα από τους δε και να κάνουμε την Ευρώπη και τον κόσμο να μάθουν ότι ένα μέρος με περισσότερη ισότητα μπορεί να δημιουργηθεί. Ένας χώρος που θα ζήσουμε όλη την εμπειρία του. Εσείς ως ε, εκλεγμένες αντιπρόσωποι πιστεύω ότι θα τηρήσετε την προτεραιότητα της ισότητας των φίλων στη δουλειά σας ε, σε πρώτη θέση και θα προασπίζεστε πάντοτε ακριβώ την ισότητα των δύο φίλων ανδρών και γυναικών. Σα εύχομαι καλή Παγκόσμια Μέρα των γυναικών, καθώ και ένα επικοδομητικό παραγωγικό ε, σεμινάριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. θέλουμε να σας ε, ευχαριστήσουμε για την πρωτοβουλία βάσης της οποίας το 2017 είναι το έτος αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων εδώ σήμερα. Θέλω να προσκαλέσω όλους σας να, και όλες σας να συνενώσετε τις δυνάμεις σας για να αγωνιστούμε για αυτό το στόχο. Η κύρωση της ε, σύμβασης τη Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ σημαντική. 14 κατημέλια ακόμα δεν έχουν κυρώσει αυτή τη σύμβαση περιμένουμε το τέλος Απριλίου να έρθει ένα πακέτο για την συμφιλίωση κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής και επίσης για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των και γυναικών στον εργασιακό χώρο. Συνεχίζουμε τώρα και έχω μεγάλη χαρά που μπορώ <clears throat> να χαιρετήσω εξαίρετες γυναίκες. Έχουμε ειδικούς, ειδικές καλεσμένους εφέτος και έχουν ε, αποδεχτεί τις ε, προσκλήσεις μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την κυρία Μικαέλ Ζων, η οποία είναι Γενική Γραμματεύς της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας. Η Μισελ Ζων έχει ξεφύγει από το δικτατορικό καθεστώς της ΑΙΤ και ήρθε ως πρόσφυγας στο Καναδά, όπου στο Κεμπέκ εργάστηκε ενεργά για να προστατεύσει γυναίκες οι οποίες ήταν θύματα βίας και δημιούργησε ένα δίκτυο και μετά έγινε μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος και κινηματογραφίστρια και στη συνέχεια έγινε γενική κυβερνήτης του Καναδά. Έχετε το λόγο κυρία Ζώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, υποδοχή, τη θερμή υποδοχή που μου έχετε επιφυλάξει. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποδοχή που μου επιφυλάξετε και θέλω να χαιρετήσω τα ιδιαίτερα στεναρά και πάρα πολύ σαφή σας λόγια για τα δικαιώματα της γυναικός, των γυναικών και για τη θέση των γυναικών στον κόσμο κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων, Σας χαιρετίζω επίσης. Αγαπητοί Ευρωπαίοι Βουλευτές, κυρία Επίτροπε Γιούροβα, κύριοι Πρεσβευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι είναι μια μεγάλη χαρά για μένα για είμαι <clears throat> μαζί σας με όλους, όλες αυτές και όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ, όλοι αυτοί που εμείς όπως η οργάνωση της Γαλλοφωνίας υποστηρίζουμε την γλωσσία ως μια προσέγγιση που επιτρέπει σε όλους την πολιτιστική και γλωσσική τους έκφραση. Η σημερινή ε, εκδήλωση είναι μια εκδήλωση πραγματικής διεθνούς δημοκρατίας. Για το σημαντικό θέμα το οποίο μας φέρνει κοντά σήμερα, Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω σκέφτομαι όλες αυτές τις γυναίκες και όλα αυτά τα κορίτσια που συναντώ σε όλες τις χώρες που πηγαίνω στις πέντε υπήρους του κόσμου και πρόσφατα ήμουνα στο Τσιπούτι, στον Ήγηρα πέρασα από το Μπουρκίνο, Μπουρκίνα Φάσο Και έχω ακόμα στο μυαλό μου τις μαρτυρίες τους, τις εξομολογήσεις γυναικών και κοριτσιών για την κατάσταση, την πολύ συχνά δραματική και αφόρητη κατάσταση που ζουν, βίας και αδικίας. <clears throat> τα καθημερινά βασανιστήρια που αντιμετωπίζουν και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, αλλά θυμάμαι και την γενοδορία τους, την αγωνιστικότητά τους, το γεγονό ότι κάθε μέρα επενδύουν στον αγώνα αυτό για να μπορέσουν να δράσουν σε όλες αυτές τις ε, συνθήκες και να υπάρξει αλλαγή. Είναι πάντα εντυπωσιακό το να μπορούμε να δούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει παρά τα εμπόδια που είχαμε. Οι γυναίκες παράγουν, οι γυναίκες καινοτομούν, οι γυναίκες αγωνίζονται, οι γυναίκες επενδύουν τις προσπάθειές τους πλήρως. Χρησιμοποιούν όλο το είναι τους, όλη την ενέργειά τους, τη δύναμή τους για να αλλάζουν τα πράγματα. Είναι σημαντική η συνεισφορά τους και πολλές φορές δυστυχώς υποτιμάται ο, λόγος, ο ρόλος των γυναικών, ακόμα και αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση. εμείς ως γυναίκες <clears throat> γνωρίζουμε ποιο είναι ο αγώνα των γυναικών σε όλα τα μέρη του κόσμου. Σε μερικές περιοχέ του κόσμου αυτό είναι ακόμα πιο έντονο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει να βγούμε από το βασίλειο της σκιά. Πρέπει οι γυναίκες να βγουν από την κρίζα ζώνη. Πρέπει να βγουν από τους νεφελώδεις αυτούς χώρους όπου παραμένουν αόρατες και δεν έχουν καμία αναγνώριση, καμία υποστήριξη στον κοινωνικό τομέα. 80% των ατόμων που εργάζονται στην κρίζα οικονομία είναι γυναίκες. Πρέπει να πράξουμε λοιπόν τα πάντα για να δοθεί μια δίκαιη αμοιβή στο έργο αυτών των γυναικών. Γιατί αυτές οι γυναίκες ουσιαστικά καλύπτουν όλη την οικιακή σχεδόν εργασία στον κόσμο. Αυτές οι γυναίκες που καταβάλουν τόσες πολλές ε, προσπάθειες φέρουν στους ώμους τους <clears throat> την Αφρική, τις χώρες του Ινδικού ωκεανού, και του Ειρηνικού ωκεανού. Και το ίδιο και στην ίδια την Ευρώπη. Μπορεί να είναι εργάτριες, μπορεί να είναι γεωργοί, μπορεί να είναι καλλιτέχνητες, μπορεί να είναι επιχειρηματίες. Με τις προσπάθειές τους μπορούν να κρατήσουν τον οικοκυριό τους αλλά και την κοινότητά τους σε ζωή. Πολλές φορές είναι μόνες τους, βασίζονται μονάχα στο δικό τους θάρρος, στη δική τους στεναρότητα, στη δική τους επιμονή. Γιατί ακόμα στον 21ο 21ο αιώνα πολλές φορές οι γυναίκες στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση ούτε στην ιδιοκτησία, ούτε στην άμεση χρηματοδότηση, ούτε σε όλα αυτά τα οποία θα ήταν απαραίτητα για να μπορέσει να εδραιωθεί ο ρόλος του στο εμπόριο, στην αηφόρο ανάπτυξη, γενικά στον οικονομικό στίβο. Και παρόλα αυτά όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι η παγκόσμια ευμάρεια βρίσκεται στα χέρια των γυναικών. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς τώρα να ανεχόμαστε το γεγονός ότι τόσα κορίτσια στον κόσμο δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε στο σχολείο και δεν μπορούν στη συνέχεια να έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανώτατη εκπαίδευση, ούτε καν επαγγελματική. Αυτές οι διακρίσεις, <clears throat> αυτές πολλές φορές καθορίζουν το μέλλον των κοριτσιών αυτών από την εποχή που είναι παιδιά και έφηβες, δηλαδή όταν παντρεύονται ακόμα και πριν από τα 16 τους. Αυτές οι διακρίσεις πολλές φορές δείχνουν μερικές φορές να υπάρχει και μία υπαναχώρηση στις κατακτήσεις των γυναικών που πολλές φορές διαρκεί γενιές ολόκληρες γυναικών. Βλέπουμε να ενισχύονται πολλές φορές τα σεξιστικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις κατά των γυναικών. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια στεναρή πολιτική θέληση για να περάσουμε ήδη από τώρα από τα λόγια στις ε, πράξεις, γιατί τα λόγια είναι πολύ εύκολα, αλλά χρειάζεται μια πολιτική θέληση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες πράξεις. Χωρίς αυτή τη θέληση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών. Σε όλους τους θεσμούς, σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υπάρξει το σπάσιμο των στερεοτύπων <clears throat> και η αλλαγή της νοοτροπίας. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεκριμενοποιήσουμε τους στόχους αυτούς, γιατί δεν έχουμε σε 22 χρόνια ακόμα καταφέρει να επιτύχουμε τους στόχους του Πεκίνου, δηλαδή τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Πιστεύω ότι όλες μας πρέπει να συνεχίσουμε όπως και στο παρελθόν να συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να αντιμετωπίσουμε τις προκαταλήψεις και τις αρνητικές νοοτροπίες, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας για να αναπτύξουμε το ταλέντο μας και τις ικανότητές μας που είναι απαραίτητα σε όλες τις χώρες του κόσμου και που πολλοί θεωρούν να τα κρατήσουν αποκλειστική ιδιοκτησία των ανδρών. Δεν έχουμε πια χρόνο να χάσουμε. Δεν έχουμε το χρόνο να χάσουμε το χρόνο μας. Σε μια στιγμή που μας λένε ορισμένοι ότι το, το status quo αποτελεί ήδη πρόοδο. πρόοδο. Όταν γίνονται νομοθετικές προσπάθειες για να υποχωρήσουν τα δικαιώματα των γυναικών, αυτά που είναι ήδη κεκτημένα, τότε πρέπει εμείς γυναίκες αλλά και άντρες θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δράσουμε <clears throat> όλοι μαζί σε όλα τα μέτωπα και γνωρίζοντας πόσο κατεπίγουσα είναι αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να διατηρήσουμε την απαραίτητη επαγρύπνησή μας και να ξέρουμε ότι είναι πράγματι απαραίτητο να αλλάξουν τα πράγματα. Απευθύνομαι λοιπόν σε εσά, πιστεύω ειλικρινά ότι η ευφυΐα ενός ανθρώπου, ενός άνδρα, καταδεικνύεται και από τη θέλησή του να προσεγγίσει τις γυναίκες και να αγωνιστεί μαζί τους. Γιατί το αντίθετο είναι μία ανοησία, μία βλακεία, μία έλλειψη λογικής. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπερασπιστεί κανένας. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρία ε, Πρόεδρε της Επιτροπής Ισότητας των Φίλων για αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει και που υποστηρίζουμε όλοι και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου απευθύνεται αυτήν την πρόσκληση να λάβω το λόγο ως Γενική Γραμματέας της Γαλλοφωνίας ενώπιον αυτής της διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης. και είναι ακόμα ένα δείγμα της εταιρικής σχέσης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διεθνούς Οργάνωσης της Γαλλοφωνίας, μιας εταιρικής σχέσης, που θα ενισχυθεί και από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράψαμε στη Μαδαγασκάρη πέρσι το Νοέμβριο στο περιθώριο της Συνόδου των Αρχηγών Κρατών και Κυβέρνησης της Γαλλοφωνίας. Είμαστε τώρα 84 κράτη σε 5 υπήρους. Είμαι λοιπόν εδώ παρούσα για να σας πω ότι ο φορέας μα είναι ε, πεπισμένο ότι πρέπει να ενώσει τι δυνάμει του μαζί σα, ώστε όλοι μαζί, τοπικέ περιφερειακέ κυβερνήσει, εθνικέ κυβερνήσει, ευρωπαϊκοί θεσμοί, κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να δράσουμε για να μπορέσουμε να θέσουμε τέρμα στι παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι τόσο συχνά και θύματά τους για να σταματήσουν Η διακρίση στην πρόσβαση στην εργασία και στην παιδεία, στην προστασία στα κοινωνικά θέματα, στου παραγωγικού πόρου και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάση σε όλου του τομεί. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε την ισοτιμία σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα, στερεότυπα, σε σχέση με το ρόλο των φίλων, που δυσκολεύουν τη ζωή όλων μας ακόμα και στις κοινωνίες όπου έχει υπάρξει κάποια πρόοδο σε σχέση με την ισότητα των φύλων. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η κοινωνικό πολιτιστική επανάσταση, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν αυτά τα μέτρα που θα επιτρέψουν σε όλα τα κορίτσια με ασφάλεια να έχουν πρόσβαση σε μια παιδεία ποιότητος. Να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα κορίτσια όχι στο όνομα αυτών που περιορίζουν το λόγο θρησκείας ή λόγω εθήμων την πρόσβαση στην παιδεία και στην αξιοπρέπεια. Θα πρέπει να στραφούμε εναντίον αυτών που αμφισβητούν την οικουμενικότητα των αξιών που έχουν να κάνουν με την ισότητα των ανδρών και των γυναικών ή που ακόμα και γνωρίζοντα αυτέ τι αξίε τι παραβιάζουν κάθε μέρα. Μπορώ να σα πω λοιπόν ότι μπορείτε να βασιστείτε στο Διεθνή Οργανισμό τη Γαλλοφωνία, κυρίω στην εμπειρία που έχουμε συλλέξει στι πέντε υπήρου του κόσμου. <clears throat> Εδώ και 20 χρόνια εμεί έχουμε κινητοποιηθεί υπέρ των ε, δικαιωμάτων των γυναικών και τη οικονομική του αυτονομία και στον αγώνα κατά τη βία που ασκείται εναντίον των γυναικών. Μέσα στα 84 κράτη μα, σε όλες τις πτυχέ τις δράσεις μας στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επίσης. Εμείς επιχειρηματολογούμε πάντα και ακολουθώντας τη χρήση της γαλλικής γλώσσας που είναι αυτό που μας ενώνει, συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Αυτό πράττουμε και σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τόνισα από την αρχή πόσο χαίρομαι για την γλωσσική πολυμορφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέραν της επιχειρηματολογίας μας και της συνηγορίας μας θέλουμε να τονίσουμε πάντα σε όλα τα προγράμματα πόσο σημαντική είναι η ισότητα ανδρών και γυναικών. Είτε πρόκειται για προγράμματα τα οποία είναι υπέρ της ειρήνης, υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, είτε πρόκειται για προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά προγράμματα, είτε πρόκειται για προγράμματα υπέρ της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, είτε πρόκειται για προγράμματα υπέρ μιας φόρου και ισοδίκαιας ανάπτυξης. Σε όλους τους τομείς λοιπόν έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες γυναικών να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και να μπορέσουν να εργαστούν από κοινού ως δίκτυο. Εδώ και δύο χρόνια στην υποσαχάρια Αφρική υποστηρίζουμε το επιχειρήν από την πλευρά των γυναικών υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ή τη δημιουργία ε, εκολαπτηρίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τομείς οι οποίοι είναι καινοτόμοι και έχουν προσθέμενη αξία. Μετά από τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε καταγάγει, νομίζω ότι έχουμε απόλυτο δίκιο που επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε αυτές τις ζωντανές δυνάμεις, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη, την δημιουργικότητα και επίσης με τον τρόπο αυτό δίνουν πραγματικά κάποια προσθέμενη αξία χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες που έχουν οδηγήσει σε μια επανάσταση στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης και μας επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες, να αλλάξουμε κλίματα παραγωγής και να ξεπεράσουμε να σπάσουμε όλα τα όρια. Εδώ θέλουμε περισσότερη ευημερία και περισσότερη, περισσότερο βιωτικό επίπεδο προ όφελο ε, των απλών ανθρώπων. Και το βλέπω και στην πράξη. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. Ε, βλέπουμε πραγματικά να δημιουργούνται νέα εργοτάξια τόπιο που μπορούμε να εργαστούμε με ελπίδα σε χώρες, σε μέρη που ε, φαίνεται να τις έχουν καταλήψει πρόοδος και ευημερία. Οι γυναίκες ε, ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για όλα αυτά και οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν και όλα αυτά μας δικαιώνουν. Οι μελέτες του ΩΣΑ του Διεθνούς Ομασματικού Ταμείου, όλο, όλα τα λένε να ε, επενδύσετε στην οικονομική δραστηριότητα των γυναικών, των νέων, να βγουν από την άτυπη εργασία, από την παράνομη εργασία. Θα δείτε αμέσως τον αντίκτυπο στην ε, ανάπτυξη, την ανάπτυξη που είναι συμμετεχική, στην ανθρώπινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σίγουρο ότι θα επηρεαστούν οι οικονομίες και τα ΕΠ όλων των χωρών. Το να μην το κάνει κανείς δεν έχει νόημα, δεν έχει λογική. Εδώ όσοι διστάζουν να επενδύσουν στις οικονομικές πρωτοβουλίες των γυναικών λέγοντας είναι επικίνδυνο, πω, πω, μπορεί να μην τα καταφέρουν, όχι. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να μην το κάνουν όταν δεν το κάνουμε αυτό, τότε υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, διότι τότε φρενάρεται η σταθερότητα, τότε ε, μπλοκάρεται η σταθερότητα για τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι ο ρόλος ο δικός σας, ο ρόλος σας είναι καθοριστική σημασίας. Ένα από τα προνόμια και τις αρμοδιότητές μας, αρμοδιότητές είναι η έγκριση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ξέρω ότι θα κινητοποιηθείτε ε, ε, αόκνος ώστε η ισότητα ανδρών και γυναικών συστηματικά να υλοποιούνται σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης. Έχω κατεξοχήν υπόψη το εργαλείο χρηματοδότησης ε, για την ανάπτυξη. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πια χρόνο. Δεν έχουμε πια χρόνο να χασομεράμε. Ο στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι υλοποιήσιμος και εφικτός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μικέλ Ζω. Είπατε πόσο σημαντικό είναι να ξεπερνούμε τα στερεότυπα. Ότι χρειάζεται βούληση και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Ταγιάννη που ήρθε κοντά μας πρέπει να αποχωρήσει γιατί έχει μια άλλη εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Μέλη κολέγος, μέλη μου συστηκήμα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι βουλευτές. Συνεχίζουμε την εκδήλωσή μας και θέλω να σας παρουσιάσω την επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Βαντάνα η οποία είναι συγγραφέας και αγωνίστρια, οικονομική σύμβουλος, μητέρα από την Ινδία. Είναι φυσικός, είναι αγωνίστρια για τα κοινωνικά δικαιώματα, έχει κάνει αγώνες για την οικολογία. για το περιβάλλον, για το ε, εμπόριο σε έντιμους όρους, για την αηφόρο γεωργία αγωνίζεται κυρίως με τις γυναίκες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Έχετε το λόγο. Cool. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και εύχομαι πολύ πολύ καλή ημέρα των γυναικών. Και όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για όλους. Ιδιαίτερος για όλους τους άντρες. Ώστε να είμαστε όλοι πιο θηλυκή. Αυτό που ο Γκάντι έλεγε ότι σημαίνει άνθρωποι με περισσότερη ενσυναίσθηση. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε όχι με ένα βιολογικό χαρακτηριστικό, όχι με ένα εγγενές χαρακτηριστικό, αλλά με ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό. Αυτό διδάσκει και η κοινωνία ε, ότι δείχνουν οι γυναίκες την συνέστηση και βέβαια αυτή βοηθά στην ειρήνη, όπως αντίστοιχα το μίσο βοηθά τον πόλεμο. Για να δούμε λοιπόν, χειραφέτηση τη γυναίκα και οικονομία. Η οικονομία που απορρέει από τη λέξη οίκο. Την ίδια λέξη από την οποία απορρέει και η λέξη οικολογία. Τι σημαίνει οίκο, οικονομία. Διαχειρίζομαι τα του οίκου μου. Κάνω να, να τρέχει το σπίτι. Το ίδιο και ο κόσμος, η οικολογία, η υφήλιος, η οικολογία λοιπόν η διαχείριση τη υφηλίου. Οι γυναίκε ήταν, είναι και θα είναι και στο μέλλον η βάση τη πραγματική οικονομία. Χτίσαμε όμως, δημιουργήσαμε άλλες οικονομίες, οι οποίες είναι οικονομίες γυναικών, είναι τυφλές μάλλον στις οικονομίες των γυναικών, στις οικονομίες της φύσης. Στοιχεία δεν θα σας δώσω γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο. Είναι προφανή όμως τα στοιχεία. Η μεγαλύτερη οικονομία είναι η φύση η δεύτερη μεγαλύτερη η γυναίκα, η γυναικεία οικονομία. Και υπήρξε και μια λεγόμενη οικονομία της αγοράς. Όταν όμως 8 άντρες ελέγχουν το ίμιση του πλούτου κόσμου, δεν βλέπω σε τι μπορεί αυτό να φέρει ισορροπία. Το 2010 είχαμε 388 δισεκατομμυρίουχους που έλεγχαν το μισό πλούτο του κόσμου. 177 ήταν το 2011, 159 το 2012. Πέρσι 62. Πάλι πολύ λίγοι. Φέτο είναι 8 αυτοί που ελέγχουν το 5% του παγκόσμιου πλούτου. Με τέτοιε τάσει λοιπόν πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ισότητα σε ένα σύστημα το οποίο είναι εκ τη φύσεω τόσο άνισο που βγάζει στο περιθώριο όλο και περισσότερους ανθρώπους και βέβαια κατά τη διαδικασία αυτή οδηγεί και σε όλο μεγαλύτερη βία. Η οικολογία και η οικονομία απορρέουν από την ίδια ρίζα και εγώ προσωπικώς δεν θέλω οικολογία σε ένα νεκρό πλανήτη, γιατί προς τα εκεί πάμε, τρέχοντας. Αν κοιτάξουμε τις κλιματικές αλλαγές, αν κοιτάξουμε την απερίμωση, την κρίση σχετική με το νερό, τα προβλήματα που επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα εκφράζει η πορεία των γυναικών για το νερό. Ήμουνα ε, σε μια διεθνή οργάνωση ε, για την ε, γυναίκα. Μετρήσαμε ε, πολλά εκατομμύρια ημερών της γυναίκας, ε, πορείας δηλαδή των γυναικών για να βρουν νερό, για να αγωνιστούν κατά τον ε, δηλητηριασμένο νερό. Η Κάρσεν πριν από 52 χρόνια έγραψε το τη σιωπηλή προσευχή. Οι γυναίκες πριν από, 40 χρόνια, ε, πριν από 30 χρόνια όρθωσαν τον άστημα κατά της μόλυνσης του Τσερνομπίλ. Στη δική μου την πατρίδα επίσης ξεκινήσαμε τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος με τη χειραφέτηση της γυναίκας. Η εξουσία, οι γυναίκες και η εξουσία. Όλοι θεωρούμε ότι την εξουσία θα μας τη δώσει κάποιος άλλος. Μα η ανδροκρατούμενη εξουσία είναι εξουσία κυριαρχίας. Όμως εμείς μιλούμε για εξουσία δημιουργική και μη βιαή. Στη δική μου την ε, κουλτούρα έχουμε μια λέξη για αυτή την ε, κουλτούρα της εξουσίας της γυναίκας που δεν είναι βίαιη. Σάκτη λέγεται. Σημαίνει αρμονία με το σύμπαν. Και είμαστε ισχυρές, το βλέπουμε κάθε φορά και μάλιστα σε περιόδους μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, η ηγεσία των γυναικών, αυτό το λίγο φως, το αμυδρό φως που μας δείχνει ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχουν θέματα πραγματικού πλούτου που σήμαινε τι. Το να είμαστε καλά. Ευημερία σημαίνει το να είμαστε καλά, όχι το να έχουμε πολλά λεφτά. Το well-being, ευημερία, σημαίνει ότι ε, περνάμε καλές ημέρες. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Ας συνεχίσουμε. Και ας συνεχίσουμε παρά τις αντίξωες, παρά την απόγνωση, με όλα τα προγράμματα της λιτότητας, τις δυσκολίες, που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τι γυναίκε που πάνε να δουλέψουν σε πέντε και 6 διαφορετικέ θέσει εργασία για να ζήσουν τι οικογένειε του και τι κοινότητε του. Πρέπει λοιπόν πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να απαλλαγούμε από τι διαδικασίε τη υποταγή των γυναικών. Μέχρι να το κάνουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτρέψουμε στις γυναίκες να ασκήσουν την ισχύ τους, την εξουσία τους. Και θα δούμε τότε ποια είναι η συμβολή τους με την γνώση τους, με την παραγωγικότητά τους. Η περισσότερη δουλειά που έχω κάνει τα τελευταία 50 χρόνια ήταν να μετρώ παραγωγικότητα και γνώση. Στοιχεία. Πλασματικά ε, δεδομένα και όρια πλούτου που τεχνητά δημιουργήθηκαν. Δηλαδή ότι αν κανείς δεν καταναλώνει αυτά τα οποία, δεν παράγει αυτά που καταναλώνει, τότε δεν μπορεί να ζήσει. Αυτό είναι το όριο για να μπορέσει να εξαπλωθεί ο πόλεμος. Μα αυτό που κάνουν οι γυναίκες, παράγουν αυτό που καταναλώνουν, δουλεύουν στα χωράφια, βάζουν φαγητό πάνω στο τραπέζι. 75% της ε, οικονομίας των τροφίμων το διαχειρίζονται οι γυναίκες. 100% στους σπόρους, γιατί εγώ δουλεύω ιδιαίτερα στον τομέα των σπόρων, περνάει από τα χέρια των γυναικών. Αν και πολλοί προσπαθούν να πάρουν αυτή την οικονομία από τα χέρια των γυναικών. Δεν θα τους επιτρέψουμε όμως. Συνεργάζομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία εις βάρος της Ανίνα Μπάσμα Θιαράης. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Μερικές φορές ε, ξεκινούμε με δεδομένο ότι οι γυναίκες είναι ανίδεες, ότι δεν ξέρουν. Όχι, όμως έχω κάνει εγώ μελέτη και μάλιστα δακτορική διατριβή για την τοπική γνώση και την μετάδοση της. Αυτή είναι η δουλειά που βλέπω εγώ ως πρόσφορα της γυναίκας και παραγωγικότητα και δημιουργικότητα που πρέπει επιτέλους να αναγνωριστούν. Εν τέλει, να δρούμε μαζί. Δεν μπορούμε αυτό να το δούμε σαν ένα είδος πατερναλιστικής προσέγγισης. Δρούμε μαζί σημαίνει βαθύ σεβασμό, βαθία ισότητα. Δρούμε μαζί σημαίνει δουλεύουμε για το κοινό καλό. Δουλεύουμε, δρούμε μαζί σημαίνει έχουμε κοινούς στόχους. Ε, με τον πλούτο που μας έχει προσφέρει η φύση, τα δάση μας, τους ποταμούς, μας, τους τη φύση, η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ρήπανση είναι αυτή η οποία κλείνει, βάζει φραγμούς και στο παγκόσμιο εμπόρεγο, γιατί αυτοί οι ολίγοι που ρηπαίνουν προξενούν και τα προβλήματα στις συναλλαγές τις εμπορικές. Έχουμε γυναίκες που δουλεύουν χωρίς μισθούς. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνίες βιώσιμες με τους όρους αυτούς. Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν σημαίνει ακόμη έναν φραγμό, μια σειρά από φραγμούς και φράκτες. Και εν τέλει ο αγώνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο στόχος της δημοκρατίας κινδυνεύει. Κινδυνεύει σοβαρά. Δρούμε μαζί λοιπόν και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την κοινή δημοκρατία, όχι την δημοκρατία των προνομιούχων. Η κοινή δημοκρατία του κοινού ανθρώπου είναι η δημοκρατία της γης, όλων των πλασμάτων. Έτσι τη λέω εγώ, δημοκρατία της γης. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τον πατριαρχικό ε, μύθο ότι είναι νεκρά ύλη η φύση ύλη προς εκμετάλλευση, ενώ έχουμε 300 τόσα δισεκατομμύρια είδη που ζουν πάνω στον πλανήτη. Εγώ δουλεύω πολύ με τα τρόφιμα ε, και βλέπω ότι την ευφυΐα με την οποία τα βακτηρία δουλεύουν μέσα στο έντερό μας, από αυτά έχουμε να διδαχτούμε. Έχει πολλά να μας δείξει ακόμα η ε, επιστήμη. Οι μικροοργανισμοί που αναζωογονούν το χώμα είναι κάτι από το οποίο πρέπει να διδαχτούμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε να ε, φωνευτεί ένας πλανήτης ζών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει με εκμετάλλευση της φύσης της γυναίκας, της φύσης της γυναίκας και των πιο αδύναμων. Πρέπει λοιπόν τώρα να δείξουμε περισσότερη ανθρωπιά ως μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, της οικογένειας του ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μάλιστα καμιά χάρη στις γυναίκες. Εγώ δεν το βλέπω έτσι το πράγμα. Σε, αυτό σε αυτή τη φάση της ιστορικής εξέλιξης, όπου θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα στάδιο ζωής στο μέλλον, που δεν θα είχε ε, το δικό μας το ανθρώπινο είδος μέλλον στον πλανήτη, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας έχει μπει στο περιθώριο, που μόνο με τη βία μπορεί να επιβιώσει. Για κοιτάξτε τι συμβαίνει στο Μεξικό. Μετά την καταστροφή, την καταστροφή της οικονομίας του ολόκληρης, το 1 τρίτο της οικονομίας του Μεξικού. στηρίζεται στα ναρκωτικά το έγκλημα της απαγωγές εις βάρος γυναικών. Κοίταξα τη δική μου την πατρίδα επίσης, πώς έχει ενισχυθεί η βία μεταξύ των ανδρών και ε, αυτό ο ενισχύεται όσο οι κοινέ βάσεις μιας κοινωνίας συνθλίβονται και συμπιέζονται. Άρα λοιπόν οι γυναίκε πρέπει να λάβουν ένα νέο ηγετικό ρόλο. Όχι να διεκδικήσουν να διώξουν του άντρε έξω, αλλά να διεκδικήσουν ένα ρόλο ηγετικό, όχι για να είναι οι ίδιε οι ηγέτε, αλλά για να υπάρχει ηγετικό ρόλο για τη μία ανθρωπότητα σε αυτόν τον ένα πλανήτη. Οι γυναίκες έχουν το δυναμικό. Για να έχουμε ένα μέλλον γυναικείο, αν έχουμε ένα μέλλον γυναικείο θα έχουμε και μέλλον ως ανθρώπινο είδος. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, ως είδος ο άνθρωπος δεν θα έχει μέλλον σε αυτόν τον όμορφο υπέροχο πλανήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρ Σίβα. Ορθά είπατε ότι η γνώση και η δημιουργικότητα των γυναικών είναι απεριόριστη. Αυτό είναι αλήθεια. Και σας ευχαριστώ. Είδατε ότι υπήρξε θερμό χειροκρότημα στο τέλος της ομιλίας σας, γιατί το μήνυμα που στέλνετε είναι τόσο σημαντικό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην, κυρία Αλία Ελ που είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Περιφερειακό Γραφείο του ΟΗΕ για την Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Ο Οργανισμό των Εθνών είναι ένα από του πιο στενού εταίρου μα, ιδίω για το σημερινό γεγονό. Έχετε το λόγο, κυρία. Εξοχότατε, κυρία Πρόεδρε, εξοχότατε, κυρία ε, Επίτροπε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίε και κύριοι. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των Γυναικών. Οι γυναίκε των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίσουν την ευκαιρία αυτή να είναι μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση η οποία συνδέεται τόσο πολύ με τις άλλες εκδηλώσει εορτασμού που λαμβάνουν χώρα στο όλο τον πλανήτη μας για την Διεθνή ημέρα των Γυναικών με το κεντρικό θέμα ο αλλάζον χώρο εργασία και η επίτευξη ενό πλανήτη 50-50 μέχρι το 2030. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επίση προσκάλεσε κοινοβουλευτικού από όλο τον κόσμο σε αυτή τη σημαντική συζήτηση για την δυνατότητα χειραφέτηση των γυναικών. Θυμόμαστε όλοι κάθε χρόνο πόσο μεγάλη πρόοδο έχει επιτευχθεί από τότε που ξεκίνησε η πρώτη ημέρα των γυναικών στη Νέα Υόρκη το 1999 για να τιμήσει τις γυναίκες που κατέβηκαν σε παιδιά για καλύτερες ε, συνθήκες εργασίας και στη συνέχεια <clears throat> η μέρα των γυναικών την χάνει εορτασμού από το 1911 από πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπου στην Αυστρία, Γερμανία, Δανία και Ελβετία. Ήταν μια ευκαιρία να δώσουμε δικαιώματα στι γυναίκες, το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγονται, να έχουν αξιοπρεπή εργασία, να παίρνουν μια αξιοπρεπή αμοιβή, να ζουν με αξιοπρέπεια τη ζωή του. Και είμαστε σήμερα εδώ λόγω του ε, συνεχούς αγώνα γενναίων γυναικών και των ανδρών που μας βοήθησαν και μας υποστήριξαν στον δρόμο αυτό για την ισότητα. Πάνω από ένα αιώνα αργότερα, πολλές από τις διεκδικήσεις αυτών των γυναικών έχουν γίνει πραγματικότητα και χάρη σε αυτές τις γυναίκες είστε σήμερα κάποιες από εσά ως κοινοβουλευτικοί. Αλλά όσο εμείς γιορτάζουμε αυτέ τι ε, επιτυχίε και τι κατακτήσει και θέλουμε να τι διατηρήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μα πάρα πολλέ προκλήσει, αδικία, ανισότητα και έλλειψη ασφάλεια. Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλε ανισότητε σε επίπεδο φύλου στην οικονομική ζωή. Οι γυναίκε κάνουν το 52% τη συνολική εργασία στον κόσμο. Αλλά ενώ δουλεύουν πιο πολλέ ώρε από του άνδρε, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και χαμηλότερη ιδιοκτησία στοιχείων ενεργητικού. Υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην κάλυψη από την κοινωνική ασφάλεια και οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να είναι σε ένδια όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία. Δεν είναι εκπληκτικό λοιπόν που το βασικό θέμα για την, ε, για την Παγκόσμια ημέρα των Γυναικών είναι οι γυναίκες στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας με στόχο τον πλανήτη 50-50 μέχρι το 2030 που είναι και το θέμα που θα απασχολήσει την 61η Σύνοδο της Επιτροπής για το καθεστώς των γυναικών που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Έχουμε τους στόχους της ε, αηφόρο ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από το 2015 στον ΟΗΕ. Οι στόχοι αυτοί αναφέρουν ε, τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030 για τις γυναίκες ώστε να υπάρξει ουσιαστική ισότητα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Έχουμε επίσης το κατευθυντήριο πλαίσιο των συμπερασμάτων τη ε, Επιτροπής για το Καθεστώ των Γυναικών που υποστηρίζεται από την έκθεση που έχει τίτλο Leave No One Behind, μην αφήσουμε καμία πίσω, που δημοσιεύθηκε από το πάνελ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Αυτό το πάνελ, το πρώτο του είδου του, δημιουργήθηκε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να μπορέσει να υπάρξει ηγετικό ρόλο και κινητοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που έχουν σαν στόχο να μειώσουν το οικονομικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων σε όλο τον κόσμο. Το πάνελ αυτό στην πρώτη μου συνεδρίαση, στην 60 συνεδρίαση της Επιτροπή για το Καθεστώ των Γυναικών, το συνεδρίασε για πρώτη φορά το 2016 το Μάρτιο. <clears throat> Έκτοτε υπάρχουν πολλές περιφερειακές συμβουλευτικέ ε, συμβουλευτικές συναντήσεις που έγιναν και περιλαμβάνεται και μια τεχνική συνάντηση συντονισμού εδώ στις Βρυξέλλες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πάνελ μας δίνει κατευθύνσεις για κέρδες δράσεις που μπορούν να αναλυθούν από κυβερνήσεις, από τον ιδιωτικό τομέα, από τον ΟΗΕ και άλλους εμπλεκομένους και επίσης κατευθυντήρες γραμμές πολιτικής ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι και οι ενδείκτε των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη. Ειδικότερα η έκθεση του πάνελ έχει εντοπίσει και 7 και κέριους ε, μοχλούς για την χειραφέτηση. Το να αντιμετωπιστούν <clears throat> οι αρνητικές ρυθμίσεις και να υπάρχουν θετικά μοντέλα ρόλου. Να υπάρξει νομική προστασία και να ανασχεθούν οι διακριτικοί νόμοι και οι κανονισμοί. Να αναγνωριστεί και να μειωθεί η απλήρωτη εργασία των γυναικών, να υπάρξουν δυνατότητες γυναίκε να έχουν οικονομικά ε, στοιχεία ενεργητικού, να αλλάξει η πολιτική των επιχειρήσεων, να υπάρχει καλύτερη δημόσια πρακτική σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του δημόσιου τομέα και να υπάρξει καλύτερη ε, εκπροσώπηση των γυναικών και τη φωνή του. Θα δημοσιεύσουμε μια δεύτερη έκθεση κατά τη διάρκεια τη επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή για τι Γυναίκε, μεταξύ των οποίων έχει εντοπιστεί η μακροοικονομική πολιτική ω ένα ακόμα κέριο μοχλό για να μπορέσουν να προωθηθούν περισσότερο οι στόχοι αυτοί. Υπάρχει παγκόσμια ανάγκη να υπάρχουν πολιτικέ δημοσιονομικέ οι οποίε να είναι ευαίσθητε στα θέματα των γυναικών ώστε να υπάρξουν δημόσιε υπηρεσίε οι οποίε αντιμετωπίζουν σωστά τα δύο φύλλα. Εμεί είμαστε έτοιμε να συνεχίσουμε τι προσπάθειε μα για τη μεταμορφωτική χρηματοδότηση και να υποστηρίξουμε ένα πλαίσιο δημοσιονομική πολιτική το οποίο θα υποστηρίξει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα και δημιουργείται μια συνένεση σε σχέση με τα πρακτέα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, οι, στόχοι, οι βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης αφορούν όλες τις χώρες του κόσμου και μπορώ να σας πω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών δεν είναι μονάχα κάτι το οποίο είναι μητελές στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου μεταξύ των άλλων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν σε σχέση με τα πρακτέα και ποιος πρέπει να τα πράξει, τώρα πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η ελπίδα μου είναι ότι αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση των συζητήσεών μα στα εργαστήρια που θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα, πώ να ενσωματώσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, πώ να κάνουμε πιο σημαντικέ και πιο αποτελεσματικέ εταιρικέ σχέσει, πώ να επιταχύνουμε την αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε. Είμαι εδώ μαζί σα εκπροσωπώντα τον φορέα UN Women, δηλαδή το Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Πρόκειται για μια περιοχή μεγάλη γεωπολιτική σημασία, όπου η δική μα προσήλωση είναι σημαντική για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της χειραφέτηση των γυναικών και αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη ανεργία και το υψηλό φόρτο εργασία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω και της χαμηλής οικονομικής ανάκαμψης και των στερεοτύπων στα θέματα του φύλου. Η εντολή μα είναι οικουμενική και εργαζόμαστε για τα θέματα τη χειραφέτηση των γυναικών στο οικονομικό επίπεδο με πολλού εταίρου και στο σύστημα του ΙΟΗΕ και εκτό αυτού και με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές εμείς θέλουμε να παίξουμε το ρόλο των συνηγόρων της ε, ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών πολιτικών ή του συντονισμού, ιδίως με στο σύστημα του ΟΗΕ και σε προγραμματικό επίπεδο σε πολλές χώρες μαζί με κυβερνήσεις και οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών και περιφερειακούς ή φορείς. Θέλω να εστιάσω στον στόχο 5,1 των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη, των στόχο βιώσιμη ανάπτυξη καλύτερα, που ζητά από όλου να εξαλείψουμε τι διακρίσει αντί όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα μέρη του κόσμου και έτσι αναγνωρίζει ότι το νομικό πλαίσιο είναι κέριο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων η οργάνωσή μας, το Young Women, εργάζεται για να υπάρξουν αλλαγές νομοθεσίες για να υπάρχει ισότιμο πεδίο σε ό,τι αφορά την οικονομική ζωή των γυναικών. Έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία μαζί με τη Διακυβερνητική Ένωση που λέγεται Ορικός Χάρτης για την ουσιαστική ισότητα το 2030 με στόχο να έχουμε παγκόσμιε εταιρικέ σχέσει ώστε να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε ή να ακυρώσουμε διακριτική νομοθεσία και όχι μόνο να εγκρίνουμε αλλά και να εφαρμόσουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα προωθήσει την ισότητα των γυναικών και τα δικαιώματά του. Πάνω από 150 χρόνια χώρε έχουν ακόμα νόμου οι οποίοι διακρίνουν εναντίον των γυναικών αρνητικά. Οικογενειακό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δίκαιο υπηκότητα και ηθαγένεια και νομοθεσία σε ό,τι αφορά την κληρονομιά, την ιδιοκτησία και τον έλεγχο τη γη και άλλων φυσικών πόρων. Μέχρι το 2030 όμω καμία χώρα δεν θα πρέπει πια να έχει τέτοιου είδου νομοθεσία κατά των γυναικών. Υποστηρίζουμε όλε τι δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με την προσπάθεια υποβοήθηση των γυναικών να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή στο ίδιο επίπεδο και με τα ίδια δικαιώματα όπω και οι άνδρε, ιδίω στι πιο φτωχέ περιοχέ και από την πλευρά των πιο φτωχών και τρωτών γυναικών. Τα προγράμματα μα έχουν σαν στόχο να βοηθήσουμε τι γυναίκε με το να αυξήσουν την προσθέμενη αξία τη εργασία του και να τι εκπαιδεύσουν πίσω για το επιχειρήν. Ε, συνεταιριστικέ οργανώσει των γυναικών και θέλουμε να βοηθήσουμε τι γυναίκε να έχουν πρόσβαση στι πιστώσει και στι αγορέ μέσω πολιτικέ οι οποίε είναι ευαίσθητε στι γυναίκε και είναι πράσινε επίση πολιτικέ και βιώσιμε στον τομέα τη υγεία. Ένα άλλο κέριο τομέα είναι η οικονομία τη μέρημνα. Ο στόχο ανα... βιώσιμη ανάπτυξη 5 θέτει σαν στόχο να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να δώσουμε την πρέπουσα αξία στην φροντίδα που γίνεται μέσω της οικιακή εργασίας, μέσω της παρουσίας και της παροχής υποδομών δημοσίων υπηρεσιών και με την πρόθεση της κοινή ευθύνη στο νοικοκυριό. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σε μια πρόταση για να υπάρξει καλύτερη ισορροπία εργασία οικογενειακή ζωή και μπορώ μονάχα να υπογραμμίσω πόσο κατεπίγουσα είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θετικό πνεύμα και τι κατάλληλε ρυθμίσει στον τόπο εργασία που να υποστηρίζουν την ισότητα για τι γυναίκε και πρέπει να σταματήσουμε μια κουλτούρα στον τόπο εργασία που επιβάλλει κυρώσει ουσιαστικά στις γυναίκες στου άντρε που χρησιμοποιούν χρόνο για να καλυψούν τι οικογενειακέ του ευθύνε. Πρέπει να κάνουμε όμω και περισσότερα πράγματα από ό,τι πρακτικέ ρυθμίσει και αλλαγή τη κουλτούρα. Τα συμπεράσματα τη 61η Συνόδου τη Επιτροπή για το Καθεστώ των Γυναικών τονίζουν την ανάγκη να δημιουργήσουμε και μια κοινωνική υποδομή μέρημνα, γιατί είναι σημαντικό το βάρο του απλήρωτου έργου των γυναικών στο σπίτι, που είναι και εμπόριο εμπόδιο στην πλήρη συμμετοχή του στην αγορά εργασία σε επίπεδο ισότητα με του άνδρε. Έχουμε λοιπόν ένα σαφέ έργο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα ήδη να εργαζόμαστε με άλλου τρόπου, νέου τρόπου για ένα καλύτερο μέλλον. Πιστεύω και προσβλέπω συζητήσει μα σε αυτή την εκδήλωση για να δούμε πώ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όπω λέει ο εκτελεστικό μα διευθυντή, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολυπλοκότητος υπάρχουν απλές αλλά σημαντικέ αλλαγέ που πρέπει να γίνουν για του άνδρε να γίνουν πραγματικοί γονείς, οι γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο και στον τόπο εργασία και οι κοπέλες να μπορούν να είναι ελεύθερες, να μεγαλώσουν ίσες με τα αγόρια. Χρειάζονται αλλαγέ από όλε τι πλευρέ αν μπορέσουμε, αν θέλουμε να έχουμε περισσότερου ανθρώπου που μπορούν να έχουν αξιοπρεπή εργασία, να παραμείνει η περιεκτικότητα για την κοινωνία αυτή και να εξασφαλίσουμε τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από όλου από την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέλη του Κοινοβουλίου, έχετε να παίξετε ένα σημαντικό ρόλο <clears throat> για να μπορέσουν να επιτευχθούν αυτές οι μεγάλες αλλαγές και να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης ώστε κανένας να μείνει πίσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που τονίσατε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει ακόμη να κάνουμε, ώστε να υπάρξει πραγματική χειραφέτηση των γυναικών. Από την πλευρά τη Επιτροπή των Γυναικών, ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε στον ε, χώρο των ίσων ευκαιριών και τη ισότητα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, όλους μας τους ομιλητές σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι ακούσαμε πραγματικά σημαντικές λαμπρές ομιλίες είναι πολύ καλή βάση για τις σημερινές μας συζητήσεις. Τώρα, για το πώς θα προχωρήσουμε. Θα χωρίσουμε το χρόνο μας σε πέντε εργαστήρια. Τα πέντε αυτά εργαστήρια θα οργανωθούν σε δύο γύρους. Τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν εγγραφεί εκ των προτέρων σε ένα από τα πέντε τα εργαστήρια θα ε, ακολουθήσουν τη συμμετοχή τους, ενώ οι ευρωβουλευτές είναι ελεύθερες και ελεύθεροι να παρακολουθήσουν όποιο εργαστήριο προτιμούν. Εύχομαι κάθε τύχη στην ε, διεξαγωγή των εργαστηρίων και να σας επισημάνω ότι μετά τη λήξη των ε, σεμιναρίων αυτών θα σας συνοδεύσουν στο εστιατόριο των βουλευτών για το δείπνο μας και αύριο θα ξαναρχίσουμε στις 9 το πρωί για να συνεχίσουμε την ε, συνάντησή μας. Στο εργαστήριο νούμερο 2 με τίτλο «Παγκόσμιες προοπτικές ελευθερία και ειρήνη και προοπτικές θα λάβει χώρα σε αυτή την αίθουσα ε, μετά από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο του εργαστηρίου αυτού, την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Τα υπόλοιπα εργαστήρια θα διοργανωθούν σε άλλες αίθουσες που μπορεί να είναι λίγο μακρύτερα. Είναι μεγάλο, μεγάλο το Ευρωκοινοβούλιο με πολλές εγκαταστάσεις και κτίρια. Θα σας, συνοδεύσει, λοιπόν, ε, θα σας συνοδεύσουν οι συνεργάτες μας που σας αναμένουν στην είσοδο. Θα σας δείξουν πώς να πάτε στις αίθουσες, οπότε σας αφήνω λίγα λεπτά για να προσανατολιστείτε και να πάτε στις αίθουσες όπου διοργανώνται τα εργαστήρια. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.